διαδικασία της Μπολόνια για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να τονίσω την ε, δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα και ιδίως το γεγονός ότι σεβάστηκε τους χρόνους της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεδρίαση έληξε. Η επόμενη συνεδρίαση θα ξεκινήσει αύριο 13 Μαρτίου από τις 9 ε, το πρωί μέχρι ε, τις 1 ε, και από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ. Μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Σας εύχομαι καληνύχτα.